και ναι, με τις αποφάσεις αυτές 2 και 7 Μαΐου. Και έτσι λοιπόν οι Μελλικές αρχές ε, όρισαν την κυρία Λίβε Τεβιρινγκ ως ε, αντικαταστάτρια του κυρίου Φίλιπ Τεμπάκερ και την καλωσορίζω και της υπενθυμίζω ότι θα πρέπει και μπορεί να, να συμμετέχει Βουλίου με πλήρη δικαιώματα και θα πρέπει να σέβεται και τις σχετικές υποχρεώσεις. Ο κύριος Μάρκος Πρέτσελ από 1η Μαΐου 2016 μπήκε στην ομάδα του ENF. Από πλευρά της ομάδας Άλτε έλαβα αιτήματα για αλλαγές ε,